Guten Morgen. Good morning. Good morning. We restart. Καλημέρα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πριν πούμε στο σημείο 43, ο κύριος Μαριάς έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Βλέπω ότι είμαι νέος βέβαια στην Επιτροπή, αλλά βλέπω για δεύτερη φορά η Γραμματεία δεν έχει συμπεριλάβει το όνομά μου στις τροπολογίες τις οποίες έχω βάλει. Διότι μαζί με τον κύριο Τσαρνιέτσκι έχω κάνει και εγώ τροπολογίες. Δηλαδή εδώ στην, α, παράγραφο, στην τροπολογία 3 έπρεπε να είναι και το όνομά μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δέστε το αυτό το θέμα γιατί μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Είμαι μεν καινούριο, αλλά να μην ε, υπάρχει η μεταχείριση αυτή γιατί έχω υπογράψει και εγώ τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. schön. Wir, wir erledigen das und äh, es ändert nichts. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε θα το κανονίσουμε. Εντάξει, μπορεί να κάνει και ένα λάθος η γραμματεία. Ευχαριστώ. Για να μην παρατείνω τη διαδικασία, θέλω να κάνω μόνο μία σύντομη παρατήρηση για τη 247 για την απαλλαγή για την Επιτροπή. Με εκπλήσει που βλέπω μια τέτοια τροπολογία, διότι θέλουμε να καταγγείλουμε παρατυπίες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο project και τελικά για να τα καλύψουμε όλα, τι κάνουμε, αναφερόμαστε σε άλλα σκάνδαλα όπως αυτό της Volkswagen και κυρίως μιλάμε για την έρευνα της Όλαφ, ε, ε, για την κυρία Λεπέν. Τι δουλειά έχει τώρα το όνομα της κυρίας Λεπέν εδώ. Είμαστε εκτός θέματος. Δεν μιλάμε για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου, αλλά για την απαλλαγή της, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρχε και μία τροπολογία που επίσης αναφερόταν στην κυρία Λεπέν και απεσύρθη και παρεμπιπτόντως να ευχαριστήσω όλους όσους την απέσυραν. πολύ κακό προηγούμενο να γίνονται αντόμινων έρευνε κατά των βουλευτών. Το 2011 θυμάστε ότι ετέθησαν να αμφιβόλω διάφοροι συναδελφοί διότι πουλούσαν τις τροπολογίες εναντί κάποιου τιμήματος και μετά ε, αρχίσαμε ονομαστικά να καταγγέλουμε αυτούς τους συναδέλφους. Ε, αν αρχίσουμε τέτοιες ιστορίες τώρα για να κρύψουμε αλλά κακό κείμενα, ε, το αποτέλεσμα θα είναι να μας κατακλείσουν τροπολογίες για άσχετες υποθέσεις ε, οι έρευνε όλα αυτέ σχετίζονται μόνο με την κυρία Λεπέν. Για δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο σχολιάζουμε μόνο την κυρία Λεπέν σε μια τροπολογία που καμία σχέση δεν έχει με το ζήτημα, αλλά σχετίζεται με την απαλλαγή τη Επιτροπή. Ναι, ευχαριστούμε. Ε, υπάρχει τεχνική διόρθωση για την Ολομέλεια. Θα βγάλουμε το όνομα και θα βάλουμε τη λειτουργία ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή να είστε σίγουρος ότι δεν θα εμφανίσετε το όνομά της. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που, λάβατε υπόψη την παρατήρηση. Μάιρες. με κυρίως Μαριάς. Ε, ε, το όνομά μου δεν εμφανίζεται και σε διάφορες άλλες τροπολογίες. Τα είπαμε ήδη με τη γραμματεία. Δηλαδή, έχω προσπογράψει διάφορε τροπολογίε και δεν εμφανίζει το όνομά μου. Μα δίνετε ένα κατάλογο με όλε τι ε, τροπολογίε που συνυπογράψατε. Ναι, ναι. Μετά τη ψηφοφορία θα έρθω σε επαφή με τη γραμματεία. Ωραία. Αρχίζουμε με το σημείο 43, απαλλαγή ο κύριος Τσέλερ είναι ο εισηγητής. Ε, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο διότι για το 2015 ε, η έκθεση για την απαλλαγή της Επιτροπής είναι συλλογικό έργο και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολλούς που συμμετείχαν, που συνέβαλαν. Το Σεπτέμβρη αρχίσαμε με την έκθεση για το ελεγκτικό συνέδριο Λάζαρο Λάζαρος. Θέλω να το τονίσω. Ήταν αγαστή συνεργασία και με τους συνεργάτες από το ελεγκτικό συνέδριο συνεχίζεται αυτή η συνεργασία με την Επίτροπο Γεωργίαβα, με τον κύριο Έτιγκαρ και το επιτελείο τους. Επίσης είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Ε, ήταν λίγα ανεπικοδομητική συνεργασία και συνεχίζουμε με τους συναδέλφους, με τον Χαν Κρίς Χινέλλας, Φίλιπ Πόρτα από τη Γραμματεία, Μπαλασέχη από την ομάδα μας και με τον Λούκας Δραέχη από το γραφείο μου. Εργαστήκαμε εντατικά για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ όλους όσους εμπλούτησαν την έκθεση με τις τροπολογίες τους, αλλά τελευταίο εξίσου σημαντικό ευχαριστώ τον Σκιώδη που μέχρι τέλος με βοήθησε με αυτή την ευρυκονομητική συνεργασία. Σίγουρα ξέχασα και κάποιους, ήταν πάρα πολλοί αυτοί που συνέβαλαν, αυτά ήταν τα κεντρικά πρόσωπα πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Ε, ναι, ευχαριστούμε. Πολύ κα... ευγενικό από πλευρά σας ε, και εμείς ευχαριστούμε του σκιώδους για τη συνεργασία και σας τον ίδιο. Περνάμε τώρα. Ε, στις 351 απολογής ε, καλύπτονται και εκτελεστικοί οργανισμοί στην απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οπότε περνάμε στο ψήφισμα, ε, περνάμε σελίδα 6 βάσει του δικού μου καταλόγου. Ε, τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται με ονομαστική απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής. Άρχεται ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Βάλτε την κάρτα σας παρακαλώ από το μηχάνημα. Είναι δύο κάρτες, αλλά δύο που δεν ψηφίζουν. Ε. Πέρασε. Χορηγείται η απαλλαγή 21 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Τώρα τροπολογία 37 για το ψήφισμα. Και κάνουμε. <laughs> Τροπολογία 37 με προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχουν ενστάσεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε παρακαλώ να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Γιατί έχει και την προφορική τροπολογία. Ε. Δεν το ξεχνάτε.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 ξέρετε ποιες θα σας πάσουν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 είναι γλωσσική διάρθρωση. 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 54, δεν ψηφίζουμε 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 58 με προφορική τροπολογία, δεν βλέπω αντιστάσει υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 με φοβολική τροπολογία δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 κατά πίπτη αυτή. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74. Όχι, όχι, στον 81 πάμε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84. Όχι. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι συμβατές, αλλά πρέπει να τις ψηφίσουμε. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ε, συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τώρα. Η επόμενη είναι 91 υπέρ. Όχι, όχι, λάθος έκανα λέει ο Με την 92 έχει προφορική τροπολογία. Ενστάσεις δεν υπάρχουν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95, απέσης, αποσύρεται, 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μόνο το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται. Όχι, έλεγχος. 97. Εγκρίθηκε 98 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ. Κατά πίπτη. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 102 δεν ψηφίζουμε. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές ελεγχός για την 104 παρακαλώ. εγκρίνεται Εγκρίθηκε. 105 ψηφίζουμε. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 107 δεν ψηφίζουμε. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 δε 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται, 122 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 123 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 124 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 125, 125 καλύπτεται. Δεν πρέπει να την ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι. 127 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος για την 127. Νομίζω εγκρίθηκε, σίγουρα δεν είμαι. Ε, the check is over. Yeah, it is adopted. Εγκρίθηκε, ναι, 128 με και τροπολογία καμία ένσταση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ. Δεν ψηφίζουμε. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133. Δεν ψηφίζουμε. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 42 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται αλλά σας παρακαλώ να ελέγξουμε καλύτερα 157 157 Πέρας. Α, ναι, απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 158 με προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω αντιρρήσει. υπέρκατα, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κρίθηκε. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές κρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 με προφορική τροπολογία, δεν υπάρχουν αντιστάσεις. υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Mm. Αποχές 183 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 92 καταπίπτει. 193 το ίδιο. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 194. Μπορούμε να ελέγξουμε για την 194 παρακαλώ. Πέρας. Α, 195 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται 196 δεν ψηφίζουμε 197 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 198 καταπίπτει 199 υπέρ 199 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται 202 <coughs> ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 203 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 210 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 211 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 213 υπέρ κατά αποχές 214 2-14 κατά πίπτη υπερ υπέρ κατά αποχές 216 2-16-17 μαζί υπέρ κατά αποχές 219 υπέρα κατά αποχές απορρίπτεται 2.18 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για την 2.18 για το 2.18 πέρας ναι εγκρίνεται 2.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.21 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 2, 22 και 23 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω εγκρίνονται τη 2 και 2, 2, 3 παρακαλώ ελέγχουμε. Απορρίπτεται. 2, 24, ε, υπέρ, κατά 2.24 παρακαλώ. Είστε όλοι υπέρ. Ε? Ξεκάθαρα εγκρίνεται. Η 2.25 καταπίπτει. 2.28. 2.28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.36 υπέρ κατά αποχές Κρίνεται. 2.37 Κατά πρώτη. 2.38 9 ε, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 2.42 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 2.43 φορική τροπολογία. Καμία ένσταση υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 2.42 44 διορθώνει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 246 υπέρ Και κατά αποχές εγκρίνεται 247 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται 247 έλεγχος Yeah, take us over. And it is adopted. Γκρίθηκε. 2.49 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.51 υπέρ. Κάτα. 2.51 λέω υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. Αλλά έλεγχος για να είμαστε και σίγουροι. 2.51. 2.51. Απορρίπτεται. 2.54. Υπέρ. Κατά. Γκρίθηκε. 2.56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.57 και 58. Ναι, όχι, 2.57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.59 υπέρ κατά α, κατά αποχές απορρίπτεται 260 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 60 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτεται 263 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτεται 264 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 271 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε 271 νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ναι. από καιρούς καιρών έχουμε ενδιαφέρουσες ε, πλούσιες. Λοιπόν, πέρας. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Συγγνώμη, λάθος. Λάθος. 2.73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πρέπει να σας πω πως η Ολλανδική καμπίνα έκλεισε, δεν υπάρχουν Ολλανδικά λόγω ασθενείας. 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 279 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη. Λοιπόν. Ωραία. Συνεχίζουμε. 2.85. 2.85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.89. Ναι να επαληθεύσουμε τη 288. 288. Πέρας. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 289. Παληθεύουμε. Κάποιοι λείπουν ακόμα. Ωραία, πέρας. Απορρίπτεται. 2,90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2,93. 2,94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνεχίζουμε 3.07 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.08 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να την επαληθεύσουμε 308. Πέρας. Εγκρίνεται. Κάποιος βάζει την κάρτα αλλά δεν ψηφίζει. Τρία δώδεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 324 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 329 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 330 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται να το επαληθεύσουμε 3.30 Πέρας απορρίπτεται 332 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία την, του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 337 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 339 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 341 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 342 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 343 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3.44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.46 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3.50 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 3.51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές απορρίπτεται, άφετ 11 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται. Δεβε 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, δεβε 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τις ψηφίσουμε όλες μαζί, 3 έως 6. Όχι. Δεβε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεβε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, DV6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, DV7 σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, DV8 σε τρία μέρη, μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή έμπλ οι πέντε πρώτες καλύπτονται από το ψήφισμα, δεν τις ψηφίζουμε, έτσι. Θέλει να ψηφίσουμε εδώ ο γραμματέας. 1 έως 5 όλες μαζί. Ναι. Όλες μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Έμπλ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Έμπλ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Έμπλ 8 μέχρι 10 μαζί. Ωραία, υπέρ. Κατά αποχέ. απορρίπτονται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. NV2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV3 υπέρ. αποχε αποχέ. απορρίπτεται. NV4 υπέρ. αποχε αποχέ. απορρίπτεται. NV5 υπέρ. αποχε αποχές εγκρίνεται. NV6 υπέρ. αποχε αποχές εγκρίνεται. NV7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε ένα μπλοκ NV10 έως 16 όχι όχι ναι πίεση λοιπόν NV10 έως 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Τρανσπορτα 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τραν 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε όλες μαζί τραν 11 ε, μέχρι 18. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ναι. Τραν 11 μέχρι 17. Ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τραν 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, τα πρώτα τρία καλύπτονται από το ψήφισμα. Να το ψηφίσουμε όλε μαζί. Ρέτζι 1 έω 3. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτονται. Ρέτζι 4 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Ρέτζι 5 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτονται. Ρέτζι 6 υπέρ. Κατά. απόχέ Απορρίπτονται. Ρέτζι 7 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. απόχέ Απορρίπτονται. Ρέτζι 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέτζι 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ρέτζι 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέτζι 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι άγκρι 1 έως 3 μπορούμε όχι Άγκρι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 3 υπέρ. Κατά. Άγκρι 3 να την επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Άγκρι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άγκρι 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 6 μέχρι 10. Μπορούμε να τις κάνουμε unblock. Όχι. Άγκρι 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 9 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 11 υπέρ κατά αποχές Να κάνουμε 12 ε, με 15 μαζί. Όχι. Άγκρι 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 14 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Δεν είναι 14 να τα πολιτεύσουμε. Κάποιοι ήταν υπέρ, κάποιοι κατά. Άγκρι 14 απορρίπτεται. Άκρη 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άκρη 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άκρη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άκρη 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άκρη 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άκρη 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πες αλληλεία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πες 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 3 έως 7 να τα κάνουμε όλα μαζί είπε κάποιος όχι 3 έως 7 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Πες 8 μέχρι 17 όλες μαζί. Πες 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, απορρίπτεται. 16 μπορούμε μαζί. 10 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Καλτ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καλτ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καλτ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλτ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλτ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καλτ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καλτ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φαμ 1 κατά υπέρ υπέρ 2 γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να κάνουμε το 3 και 4 ομού 3 και 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 5 έως 9 γυναικών μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. 21-4. Συγχαρητήρια για όλη αυτή τη δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ. Item, item 42. Το 42. Item 42, the special reports. Yeah, the special reports are now on our agenda to be voted. Σε διάταξη αυτό τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Έχετε τον κατάλογο για την ψηφορία. 2 με 10 όλες μαζί. Είναι η ειδική έκθεση του συνεδρίου. 2 με 10. Όλες μαζί συμφωνείτε. Ναι. 2 με 10. Όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Έντερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 με 22. Όχι. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά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 απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 50 με 60 όλες μαζί 50 με 60 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 με 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 73 αποσύρεται, 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά έλεγχος για το 82 Δεν είμαι σίγουρη ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πέρας απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 μέχρι και 87 όλες μαζί. 85 με 87 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτονται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ έλεγχος για το 94. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά. 95 υπέρ, κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 95. Και εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτωται. 97 υπέρ αποχή. Κατά αποχές έλεγχος για το 97. Ψηφίζομαι. And it Εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτωται. 100 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτωται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 105 Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 106 υπέρ, κατά, άποχες, έλεγχος, ίσως ίδιο το αποτέλεσμα, ίδια πλειοψηφία. Ναι, απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 107 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, ρυθμόν 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. και τώρα θα ψηφίσουμε για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε πέρας συγχαρητήρια ή για τη δουλειά σας. Το υπαριθμό 41 της σημερισίας διατάξεως όσον αφορά το Ταμείο Ανάπτυξης. Κύριο Μαρζέ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χιώδες εισηγητές που από το τέλος του παρελθόντος έτους βοήθησαν για αυτή την έκθεση. Επίσης ευχαριστώ και την κυρία Λαμάρκ από το Ελληνικό Συνέδριο, ε, την Τράπεζα Επενδύσεων, τον συνάδελφο από εκεί και τον αρμόδιο επίτροπο, τον διευθυντή της ΔΕΒΚΟ και επίσης τον ε, Διευθυντή της Υπηρεσίας για τους Πόρους αλλά επίσης και τον εισηγητή της Επιτροπής Ανάπτυξης τον συνάδελφο κύριο Ρούμπιχ, ο οποίος έχει αναλάβει την γενική έκθεση της απαλλαγής για την Επιτροπή, του κύριο Τσέλερ, τη γραμματεία της ε, Επιτροπής μας και δύο συνολικές αλλά και το σύνολο των συνεργατών μας, αλλά και πολιτικών συμβούλων. Και ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για τα ευγενικά σας λόγια προς όλους, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφοφορία. EDF. Τροπολογία παρισμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, 2. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η απόφαση χορήγησης της απαλλαγής. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζομαι. Still colleagues missing. Λείπουν κάποιοι συνάδελφοι. The, hmm? the vote is closed. 21. και συγχαρητήρια. 21-3 το σκορ. Κλείσιμο των λογαριασμών. Θα ε, χρειαστεί να ψηφίσουμε την τροπολογία 4 αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία 5 υπέρ κατά έχει εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το κλείσιμο των λογαριασμών με ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα. Still one colleague missing. Λείπει η ψήφος ενό συναδέλφου. Okay. Okay. Okay. Yeah. The vote is closed. Πέρασε. Πέρασε. 23. Και σας ευχαριστώ. Το ψήφισμα τώρα. Τροπολογία 6. Τεχνογλωσσική προσαρμογή διόρθωση. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 7. Έλεγχος. check is over and it is rejected. I'm... Απορρίπτεται. Λυπούμε. Λοιπόν, 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 9. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 11 υπέρ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 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Yeah, but I had compromise 3. Okay. Yeah, compromise 2 and 3, we had it one after the other. Compromise 4 in favor. 4, 4. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για το 44. Νομίζω εγκρίνεται. Check is ε, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 57 ήταν. 57 ήταν. Ε, έλεγχος. Πέρας. Εγκρίθηκε. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Και την 58. 26 συναδέλφους και δεν ξέρω πού είναι μέσα στην αίθουσα. Α, απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος παρακαλώ. 64. Νομίζω εγκρίνεται. Ναι, ναι, εγκρίνεται. 65 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά, αποχές, να ελέγξουμε την 67. 67. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Ωραία. Έγινε ο έλεγχος. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Έλεγχο 78. Έλεγχος 78. Πέρα εγκρίθηκε. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Ποια θέλετε, την 82. Οκ, okay, 82. Έλεγχος. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά ε, καλά, ας την ελέγξουμε και την 85 τότε καλύτερα 85 Α, μπορεί τότε Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για την 88. Για την 88. Εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 99 κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται αλλά θέλω να κάνουμε έναν έλεγχο 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 102 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι είπατε? Την 104. Καλά, να την ελέγξουμε. Ε, ΔΒ4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το ψήφισμα άρχεται. And Πέρας. 20 προς 3. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πολύ καλή δουλειά που κάνατε. Πεντατρία έως 59 τώρα. Δεν βλέπω τον εισηγητή. Α, εδώ είσαστε. Εσείς ήσασταν που λείπατε. Absolutely. Yeah. We, yes. The bio-based industries. Amendment to By BBI. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, χωρίς η απαλλαγή με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. The vote is closed. 16 προς 6. Πολύ ωραία. Κλείνουν οι λογαριασμοί. Πάμε στο ψήφισμα. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για το ψήφισμα με, την, με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 20 ψήφοι προς 3 συγχαρητήρια στον εισηγητή. Για το Clean Sky Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Για την απόφαση χορήγηση απαλλαγή. Με ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. The vote is closed. Πέρασε. Αγκρίθηκε. Κλείνουν οι λογαριασμοί. Πάμε στο ψήφισμα. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. The vote is closed. Ε, ωραία, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Excel ε, για την ηλεκτρονικά στοιχεία, δομικά στοιχεία υπέρ ε, κατά απορριχές απορρίπτεται η προτροπολογία για την χορήγηση απαλλαγής ε, νομαστική ψηφοφορία. Ναι, ναι. It is Πέρασε. This implies the closure of accounts. We go to... Κλείνουν οι λογαριασμοί. Πάμε στην τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές. Μπορούμε να κάνουμε ανέλεγχο για την ε, τροπολογία 3. The check is over and it is adopted. Amendment 4 in favor. Again. Η 5 η ε, ε, προφορική τροπολογία δεν υπάρχουν στάσει υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 αποσύρεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 αποσύρεται. Ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. The vote is closed. 20 3. Congratulations to the rapporteur. We vote on fuel cells and hydrogen. Hydrogen, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, απόφαση χορήγηση απαλλαγή με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε 19 ψήφοι προ 4. Ωραία για το ε, κλείσμα των λογαριασμών. Ε, για τη τροπολογία 7 είπαμε. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 αποσύρεται, 10 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την τροπολογία 10. Τέρμα, ο έλεγχος εγκρίνεται, ε, τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, για το σύνολο του ψηφίσματος με ψηφοφορία. Παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας. 21 προς 3. Συγχαρητήρια. Για το είναι, για τις πρωτοβουλίες, τροπολογία 1, υπερ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απόφαση χορήγηση απαλλαγής με ονομαστική ψηφοφορία. 20 προς 4 εγκρίνεται. Κλείνουν λίγο λογαριασμοί. Ε, τροπολογία 5 για το ψήφισμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, το ψήφισμα με ονομαστική. The vote is closed. And it is 21 to 3. Congratulations. 21 προς 3. Ήτερ. Νομίζω. Ε, τροπολογία 1 και 2 υπέρ. Κατά αποχές. Ε, ναι, α, ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ. Νομίζω απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Χορήγηση απαλλαγή. Ε, ονομαστική ψηφοφορία για να ψηφίσουμε για την απόφαση. Πέρα. 17 προς 7 και πάμε τώρα στο ψήφισμα για το κλείσιμο των αιτήσεων λογαριασμών. Το πολυγία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Από έλεγχος παρακαλώ για την 11. Για τη 12.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 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, ψήφισμα. Με το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. The Πέρας. <coughs> Συγχαρητήρια, εγκρίνεται. Σίζαρ. Ασφάλεια αεροπλοείας. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απόφαση απαλλαγής με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρασε. Κλείνουν και οι λογαριασμοί. Ψήφισμα τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τραν 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 αποσύρεται τραν 1 έως 7 ε, τραν 14 καλύπτεται το αρχικό κείμενο. Το ψήφισμα τίθεται σε ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρασε. 22 έναντι 3 συγχαρητήρια. Και έληξαν οι ψηφοφορίες για τις απαλλαγές. Σας ευχαριστώ για την πειθαρχία και φτάσαμε και στο τέλος της δημόσιας συνεδρίασης. Συνεχίζουμε απευθείας με συντονιστές για να γλιτώσουμε χρόνο. Τελειώνει εδώ το δημοσίο μέρος της συνεδρίασης και ε, προτείνω να συνεχίσουμε με τους συντονιστές με μια έτσι σύντομη συνεδρίαση. Everyone's free to go